Συνεχίζουμε τώρα με τις επεξηγήσεις ψήφου. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα θεσινά πρακτικά. Τα πρακτικά της ε, χθεσινής ε, συνεδρίασης και όλα τα έγγραφα τα οποία εγκρίθηκαν είναι διαθέσιμα. Έχετε αντιρρήσεις μήπως? Όχι, συνεπώς εγκρίνονται τα πρακτικά.